Αρχίζουμε λοιπόν την ψηφοφορία, το πρώτο θέμα. Κυρία Ίντφελτ, διαδικαστικό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα συνάδελφοι, ακούσαμε την, ε, το χαιρετισμό του Προέδρου της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης. Πολύ σημαντικό γεγονός. Με αυτή την ευκαιρία έχω να κάνω μια παράκληση. Πριν από λίγες μέρες ε, ακούσαμε ότι ο δόκτωρ Μουκρέγκε που βραβεύτηκε με το βραβείο Ζαχάροφ δεν θα έχει πλήρη προστασία πλέον από τα Ηνωμένα Έθνη και ένα μήνα πριν ένα συνεργάτης του δολοφονήθηκε ε, υπάρχουν απειλές κατά των συνεργατών τους και θα ήθελα η ηγεσία του Κοινοβουλίου μαζί με την κυρία Μογκερίνη που ήταν πριν από λίγο εδώ να αξιοποιήσουν όλες τις ε, διασυνδέσεις που διαθέτουν για να έχει πλήρη προστασία στο έργο που κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ λάβαμε γνώση και θα το συζητήσουμε με την κυρία Μογκερίνη, κυρία Γκόμες. I like this Και εγώ με αυτή την ευκαιρία θέλω να ζητήσω την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για να επιστήσουμε την προσοχή των μοξικανικών αρχών στη δολοφονία του Χαβιέ Πάνες Καριέρας, έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο που ε, αποκάλυψε τη διαφθορά, το τράφικινγκ και το οργανωμένο έγκλημα. Χθε δολοφονήθηκε άγρια και θα πρέπει και αυτό γίνεται για να αποθαρρυνθούν και άλλοι ερευνητέ, δημοσιογράφοι. Θα πρέπει να πούμε στι μεξικανικέ αρχέ ότι τιμούμε τη μνήμη του και ότι θέλουμε οι μεξικανικέ αρχέ να φέρουν στο δικαστήριο τους υπέτειους αυτού του αποτρόπαιου εγκλήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ελάβαμε γνώση και θα ε, προωθήσω με το έτοιμά σας. Τέλος, ε, αν μου επιτρέπετε, θα... Ε, ε, προχωρήσουμε στην ψηφοφορία ε, με τη σειρά. Πρόκειται για ηλεκτρονική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα στο, στην πρώτη έκθεση που έχετε τους πλήρες τίτλους. Ευχαριστώ. Πέρας. Ενεκρίθη. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Επόμενη έκθεση του κυρίου Πρέντα. Πάλι ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας. Εγκρίθηκε συγχαρητήρια στον κύριο Πρέντα. Η έκθεση του κυρίου Στεχόφσκι. Πάλι ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Στεχόφσκι. Βλέπω ότι είναι πολύ μετριόφρον ο εισηγητή. Δέχεται με μετριοφροσύνη τα συγχαρητήρια. Ο κύριος Ρουά, πάλι ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Α, συγγνώμη, θέλετε να λάβετε το λόγο, κύριε Ρούα. Ευχαριστώ. Πάλι θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της προσχώρησης της Ένωσης ε, στη Διεθνή Επιτροπή Βάμπακος, 27 ε, χώρες παραγωγή και καταναλωτές ε, και διαμεσολαβητές συμπεριλαμβάνονται. μέχρι τώρα δεν είχε προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στην Επιτροπή αυτή. Πρόκειται για διεθνή οργάνωση όπως αυτή που υπάρχει για το πετρέλαιο, τη ζάχαρη, το κακάο. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν είχε προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα στην, ε, στον οργανισμό αυτό. Ε, προσβλέπουμε σε, στη θετική σας ψήφο και ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ευχαριστώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Κυρία Φερχάιεν, ονομαστική ψηφοφορία και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας. εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Έκθεση Πιτέρα. Αρχίζομαι να ψηφίζω με τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται θα έλεγα. Θέλετε να γίνει έλεγχος. Καλώς. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 6 εγκρίθηκε, άρα το αρχικό κείμενο ε, μέρος 1 και μέρος 2 καταπίπτουν. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ευχαριστώ. Απορρίπτεται. 13 καταπίπτει. Α, ε, υπέρ της 13, συγγνώμη, κατά. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Επτά υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Ε, κάναμε έλεγχο. Ψηφίζομαι επί του συνόλου του ψηφίσματος. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην κυρία εισηγήτρια. Προχωρούμε. Έκθεση κυρίας Μπορζάν. Τροπολογία 2. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται ε, παράγραφος 65 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ελέγξουμε καλύτερα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Ελπίζω να μάθω γρήγορα τη διαδικασία της ψηφοφορίας. 79 υπέρ. Παράγραφος 79. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 115. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 117. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ή θέλετε να ελέγξουμε. Ας κάνουμε έναν έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίφθηκε. Παράγραφος 119, αρχικό κείμενο. Πρώτο μέρος, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη AI, τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη D, αρχικό κείμενο. Πρώτο μέρος υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Μπορζάν. Προχωρούμε έκθεση κυρίας Μπεγκίν. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Δύο λεπτά διάλειμμα για λόγους τεχνικούς. Ευχαριστώ πολύ για την βοήθειά σας ε, κατά την ψηφοφορία. Δύο λεπτά διάλειμμα και θα ξαναρχίσουμε με τις επεξηγήσεις, αιτιολογήσεις ψήφου.